Bien, por favor. Παρακαλώ. Καλώς ορίσατε. Όπως γνωρίζετε, επισήμως το δεύτερο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Το τρίτο είναι η έγκριση των πρακτικών. Και ε, μετά έχουμε τις ανακοινώσεις του Προέδρου. Επειδή όμως έχουμε εδώ τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, θα δώσουμε απευθεία το λόγο, χωρί ε, να εγκρίνουμε κάποιε αλλαγέ που έχουμε, γιατί θα πρέπει να τι συζητήσουμε αργότερα την ημερήσια διάταξη. Και περνάμε στο σημείο υπαριθμών 5 τη ημερήσια διάταξη, ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό Γεωργία ε, ε, της Ελληνικής Προεδρίας, τον κύριο Αθανάσιο Τσαφτάρη και θα περάσουμε από εκεί και πέρα στην έγκριση των πρακτικών της ημερήσιας διάταξης και των ανακοινώσεων του Προέδρου για να δώσουμε τη δυνατότητα στον ε, κύριο Υπουργό διότι σίγουρα έχει πολλή δουλειά να ε, μιλήσει εδώ σε εμά για να συνεχίσει στη συνέχεια τις εργασίες σας. Καλώς ορίσατε, κύριε Υπουργέ. Είναι χαρά μου να σας καλωσορίζω εδώ στην Επιτροπή αλληλία, Μία μικρή, μεν, αλλά σημαντική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να μας παρουσιάσετε τις προτεραιότητες της νέας ε, Προεδρίας του Συμβουλίου για το επόμενο εξάμεινο. Ε, πρόκειται για μια διαφορετική προεδρία, σου είχε ένερης, ε, διότι θα διακοπεί ε, λόγω ε, της θητείας, στη διάρκεια της θητείας σας, επειδή ακριβώς θα έχουμε τις ευρωεκλογές. Ε, βέβαια υπάρχουν αρκετά θέματα να συζητήσουμε μέχρι τότε. Ε, έχουμε τη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής, εγκρίναμε το βασικό κανονισμό, η συγγήτρια ήταν η κυρία Ρόντους, η οποία είναι εδώ μαζί μας σήμερα, δεν μπορούσε άλλωστε να είναι και αλλιώς. Και επίσης έχουμε και ε, τις εκθέσεις για την κοινή οργάνωση των αγορών. Ε, η συγγητής ήταν ο κύριος Στίβενσον για το θέμα αυτό. Ε, και τώρα έχουμε περάσει στην ουσία. Ξέρετε πολύ καλά ότι θα είστε εσείς αρμόδιος για αυτά τα θέματα, ε, την αλία των βαθέων υδάτων και ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε και συμφωνία. Εμείς από πλευρά Συμβουλίου ε, και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συζητήσαμε το θέμα, προσπαθήσαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλήξουμε σε συμφωνία. Αλλά ό,τι έγινε έγινε, θα συνεχίσουμε τώρα τις διαπραγματεύσεις, θα συνεχίσουν οι τριμερείς διάλογοι για να μπορέσουμε ίσως να ολοκληρώσουμε τα θέματα αυτά, τα οποία νομίζω ότι μας ενδιαφέρουν όλους. Ε, όλοι προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και θεωρώ ότι ε, θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Κάθε φορά που έχετε νέος προεδρεύων του λέω το ίδιο. Είναι κάτι το οποίο διεκδικούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ε, το γεγονός ότι έχουν μπλοκαρωστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό τα σχέδια διαχείρισης ε, και ε, για το γάδο υπάρχει και για άλλα είδη. Ε, έχουμε την Task Force και ελπίζω ότι και με τη βοήθεια της Ελληνικής Προεδρίας θα καταφέρουμε σε αυτή την περίπτωση να επιλύσουμε το πρόβλημα. Και υπάρχει και ένα θέμα το οποίο θα χρειαστεί να αντιμετωπίσετε κι εσείς ε, και από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντικό. Εμείς θεωρούμε ότι είναι ζωτικής σημασίας η εξωτερική διάσταση ε, της και οι εξωτερικές διαστάσεις κοινή ελευθερική πολιτική πολιτικής είναι πολύ σημαντικές. Υπήρξε μια εξαιρετική έκθεση της κυρίας Λεβίν και είναι πολύ σημαντική αυτή. Υπάρχουν κάποιες συμφωνίες οι οποίες ε, ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί, υπάρχουν και κάποιες άλλες οι οποίες πρέπει να ανανεωθούν. Για παράδειγμα, συμφωνία με τη Μαυριτανία. Υπάρχουν και άλλες όμως συμφωνίες και ελπίζω ειλικρινά ότι η Ελληνική Προεδρία θα δώσει μια σημαντική όθηση ώστε σε κάποιες περιπτώσεις να ανανεωθούν και σε κάποιες άλλες να, να περατωθούν οι συμφωνίες. Και νομίζω ότι, όπως λέω πάντα στην Προεδρία, ε, εμείς είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε, δεν είμαστε εχθρός του Συμβουλίου, ούτε εχθρός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα θέλαμε να μας βλέπετε ως φίλους που συνεργαζόμαστε από κοινού για το μέλλον του αλευτικού τομέα. Και αυτό φυσικά σημαίνει ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται πλήρως για όλα όσα συμβαίνουν και όπως προβλέπουν και οι διαδικασίες στις συνθήκες. Είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να επαναλέβω και στην Ελληνική Προεδρία. Τίποτα άλλο από πλευρά μου. Ε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ακούσουμε τις προτεραιότητές σας, τις ανησυχίες σας και από εκεί και πέρα να κάνουμε μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων με τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής μας. Ε, καλώς ορίσατε και πάλι. Και μέχρι να σταματήσει επισήμω τις εργασίες του το Κοινοβούλιο, εδώ η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Thank you. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ σήμερα με την ευκαιρία της ανάληψης της πέμπτης ελληνικής προεδρίας για να σας παρουσιάσω στην Επιτροπή σας το πρόγραμμα εργασίας στον τομέα της αλληλείας. Βρίσκομαι σήμερα εδώ για να συζητήσω μαζί σας με τον συνομοθέτη του Συμβουλίου που διαθέτει πλέον μεγαλύτερη επιρροή προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας και φυσικά προς όφελος των επαγγελματιών του κλάδου, της αλληλείας και των υδατοκαλλιεργιών. Η χρονική αυτή στιγμή Όλοι γνωρίζετε, είναι πολύ ιδιαίτερη για τη χώρα μου. Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια κρίσιμη μεταβατική περίοδο για την Ευρώπη. Σε αυτό το σημείο καμπής το μεγάλο διεκείδευμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδράζεται στην προώθηση της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης και ιδιαίτερα των νέων και της εξασφάλιση σταθερότητας και ευημερίας για όλους τους πολίτες. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει πρώτα απ' όλα να επαναβεβαιώσει την αποστολή της στην καρδιά αλλά και στο νου των Ευρωπαίων πολιτών της. Επιτρέψτε μου τώρα να αναφέρω συνοπτικά στην αρχή τις οριζόντιες προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας. Πρώτον, η τόνιση της ανάπτυξης και της απασχόλησης και της συνοχής το ένα προϋπόθεση του άλλου βασικά που μπορούν να συμβαδίσουν αρμονικά για τη δημοσιονομική με τη δημοσιονομική πειθαρχία. Δεύτερον, η στήριξη του κοινού νομίσματος και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης της κοινωνίας και των πολιτών στην ευρωπαϊκή ιδέα. Τρίτον, οι εξωτερικές προκλήσεις και η απάντηση που οφείλει να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μεταναστευτικό ζήτημα, η τραγική διάσταση του οποίου αναδεικνύεται συχνά στη θάλασσα και στα χερσαία σύνορα της Ευρώπης. Και για να περάσω στο στοιχείο της θάλασσας που χαρακτηρίζει την Ευρώπη και τη χώρα μου, η ελληνική προεδρία αναγνωρίζοντας το ζωτικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η θάλασσα στη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανάκαμψη της Ευρώπης και την κρίση καθώς και στην ανάκτηση της ανταγωνιστικότητάς της στην παγκόσμια οικονομία. Έτσι, υιοθετήσαμε μια οριζόντια προτεραιότητα η οποία διατρέχει όλες σχεδόν τις υπόλοιπες και είναι η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θαλάσσια πολιτική εκτείνεται σε τομείς όπως η αλληλεία που μας ενδιαφέρει εδώ και φυσικά τον τουρισμό μέχρι και τις μεταφορές, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας και άλλα ως προς τις προτεραιότητες στον τομέα της αλληλείας. Ερχόμενος λοιπόν στην αλληλεία θα μιλήσουμε για ένα τομέα ο οποίος όχι μόνο εξασφαλίζει εξαιρετικά ποιοτική διατρο... την εξαιρετική ποιοτική διατροφή μας αλλά συμβάλλει σημαντικά και στον σημαντικό βαθμό και στη διατήρηση του οικονομικού και κοινωνικού ιστού πολλών παράκτιων και νησιωτικών κοινοτήτων εξασφαλίζοντας την ανάπτυξή τους και μαζί με αυτήν πολλές θέσεις εργασίας σε περιοχές τις οποίες μάλιστα δεν υπάρχουν και πολλές εναλλακτικές λύσεις για ανάπτυξη και απασχόληση πέραν ίσως του τουρισμού. Τα τελευταία τρία χρόνια ερχόμενος στην μεταρρύθμιση της κοινή αλλιευτικής πολιτικής και ιδιαίτερα στο, ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Θάλασσα και την Αλληλεία τα θεσμικά όργανα δούλεψαν πολύ σκληρά ώστε να τεθεί σε εφαρμογή η νέα κοινή αλλιευτική πολιτική από την 1η του Ιανουαρίου του 2014 με στόχο τη διασφάλιση της μακροχρόνιας περιβαντολογικής, οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας του τομέα. Πολιτική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη επιτευχθεί για τον βασικό κανονισμό της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και για τον κανονισμό της κοινή οργάνωσης αγορών. Και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να σας συγχαρώ και για την εξαιρετική συνεργασία και τη συμβολή όλων σας και σας κύριε Πρόεδρε στο σημαντικό αυτό επίτευγμα. Πιστεύουμε ότι με την ίδια πολιτική βούληση θα καταφέρουμε να έχουμε παρόμοια αποτελέσματα και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας, το οποίο θα αποτελέσει την κύρια προτεραιότητα στην ελληνική Προεδρία. Είμαι πεπισμένος ότι οι συνομοθέτες έχουν την ίδια άποψη ότι το Ταμείο αυτό αποτελεί έναν από τα κύρια εργαλεία για την ομαλή μετάβαση και την υλοποίηση των στόχων μας, προκειμένου η νέα κοινή αλλιευτική πολιτική να αποδειχθεί πραγματική και να μην υπάρχουν κενά στην υποστήριξη του τομέα. Για το σκοπό αυτό είμαστε υποχρεωμένοι και πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου να καθίσουμε και πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να πετύχουμε πολιτική συμφωνία προκειμένου να εξασφαλιστεί η έναρξη ισχύω του Ταμείου το συντομότερο δυνατό. Και σε κάθε περίπτωση πριν τη διακοπή των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα μέσα Απριλίου. Είμαι βέβαιος ότι το Κοινοβούλιο συμμερίζεται αυτούς τους στόχους και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια κύριε Πρόεδρε προκειμένου η προσπάθεια αυτή να είναι επιτυχής σε ό,τι αφορά τα, πολιτικά, τα πολιετή σχέδια διαχείρισης που και εσείς αναφέρετε, υπήρξαν αιτία διαφωνίας και τριβής μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών. Η διοργανική ομάδα όμως που σχηματίστηκε, η γνωστή Task Force, βρίσκεται σε διαδικασία έβρεσης ρεαλιστικών λύσεων. Ξεκίνησε τις εργασίες της, όπως ξέρετε, την 23η Σεπτεμβρίου του 2013 συνεδρίασε ήδη πέντε φορές πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων και θα ήθελα και σε αυτό το σημείο κύριε Πρόεδρε να σας ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία και εσάς και τα μέλη του Κοινοβουλίου. Οι εργασίες έχουν ήδη ξαναρχίσει και έχουν προγραμματιστεί και οι επόμενες συναντήσεις. Οι εργασίες της Task Force επιβεβαίωσαν την καλή θέληση και των δύο πλευρών για να εξευρεθεί λύσεις. Πρόοδος έχει ήδη συμμε, σημειωθεί μέχρι στιγμής στον προσδιορισμό των βασικών στοιχείων ενός μελλοντικού σχεδίου διαχείρισης για τα λεγόμενα single stocks, τα απλά, στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και όπως γνωρίζετε η Κορεπέρ 1 ενέκρινε ήδη τα αποτελέσματα αυτά. Η Ελληνική Προεδρία θα συνεχίσει τις εργασίες της Task Force έως τον Μάρτιο του 2014 και ελπίζουμε να έχουμε περαιτέρω αποτελέσματα σε πιο σύνθετους τύπους πολιετών σχεδίων τα οποία περιλαμβάνουν και μικτούς τύπους αλληλείας. Όλοι γνωρίζουμε ότι εκκρεμεί μια δικαστική υπόθεση σχετικά με το σχέδιο για τον Γάδο, εν τούτης, βλέπουμε την ομάδα εργασίας ως μια ευκαιρία να κοιτάξουμε μπροστά ανεξάρτητα από την πολιτική διαμάχη. Και ο λόγος είναι ότι η κοινή αλλιευτική πολιτική θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό αφενός μεν από τα πολιετή αυτά σχέδια διαχείρισης και για την εφαρμογή της απαγόρευσης των απορρίψεων και αφετέρου από την περιφερειακή προσέγγιση στη διαχείριση της αλίας. Και με την ευκαιρία που ανέφερα τις απορρίψεις έρχομαι στα θέματα των απορρίψεων είναι άλλη μια προτεραιότητα που γνωρίζεται για το πρώτο εξάμεινο η οποία αφορά στις εργασίες για την εφαρμογή της απαγόρευσης των απορρίψεων όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Μόλις λάβαμε την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τις αναγκαίες τροποποιήσεις της ισχύουσα νομοθεσίας για τα μέτρα ελέγχου καθώς και για τα τεχνικά μέτρα και έχει ήδη ξεκινήσει η εξέτασή της. Πρόκειται για ένα βασικό νομοθέτημα της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και συνεπώς προτιθέμεθα να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατό με τις εργασίες αυτών των φάκελων. Σε ό,τι αφορά τα τάκ και τις ποσοστώσεις, κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 2013 το Συμβούλιο απεφάσισε, άλλωστε αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο, για τις ελιευτικές δυνατότητες, δηλαδή τα τάκ και τις ποσοστώσεις, καθώς και τα όρια αλλιευτικής προσπάθειας ανάλογα με την περίπτωση, τόσο για την Βαλτική θάλασσα, όσο και για τη Μαύρη θάλασσα, καθώς και για τις ελιευτικές ε, ευκαιρίες στα εσωτερικά και τα διεθνή ύδατα. Ωστόσο, ορισμένα από τα στοιχεία στον κύριο κανονισμό είναι προσωρινά, ένα αναμονή όπως γνωρίζετε του αποτελέσματος των διαβολεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ορβηγία και των διαβολεύσεων των παράκτιων κρατών. Συνεπώς θα απαιτηθεί τροποποίηση του κύριου κανονισμού μόλις γίνει γνωστή η έκβαση των συγκεκριμένων διαβολεύσεων. Σε ό,τι αφορά το θέμα της αλληλείας στα βαθιά ύδατα, το Συμβούλιο σκοπεύει να προωθήσει και αυτό το θέμα και τις εργασίες για την τροποποίηση του κανονισμού για την ελευθερική προσπάθεια στα βαθέα ύδατα. Ένα φάκελο αμφιλεγόμενο με δυσκολίες για το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαμόρφωσε ήδη τη θέση του. Οι συζητήσεις θα ξεκινήσουν ήδη από αυτήν την εβδομάδα. Και στο σημείο αυτό να αναφερθώ ότι θα ληφθεί δεόντως υπόψη το επικοδομητικό έργο το οποίο έχετε επιτελέσει στο Κοινοβούλιο κύριε Πρόεδρε εσείς και οι κύριοι κύριοι και οι κυρίες ε, βουλευτές. Ως προς τις ευθυγραμμίσεις με τη συνθήκη της Λισαβόνας, όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια σειρά από προτάσεις για την ευθυγράμμιση της εφιστάμενης νομοθεσίας με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε για την πρόταση εναρμόνισης των κοιτοδών και των τεχνικών μέτρων που έχουν προχωρήσει για τη Μεσόγειο και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξετάσουμε και τις άλλες προτάσεις λαμβάνοντας υπόψη φυσικά τους κοινού χρονικούς περιορισμούς που έχουμε όλοι μας. Σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική που αναφέρεται ότι είναι σημαντική για το Κοινοβούλιο σχετικά με τις αλληλευτικές συμφωνίες θα ξεκινήσουν σύντομα οι διαπραγματεύσεις για το νέο πρωτόκολλο με τη Μαυριτανία. Το τρέχον πρωτόκολλο όπως ξέρετε λύγει κατά τη διάρκεια του 2015 αλλά πιστεύω λόγω των μακροχρόνιων διαπραγματεύσεων και των διαδικασιών επικύρωσης είναι σημαντικό οι συζητήσεις αυτές να αρχίσουν νωρίς. Δεν έχουμε δηλαδή πολύ χρόνο. Επίσης θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης με τη Σενεγάλη. Οι συζητήσεις θα αρχίσουν στα τέλη αυτού του μήνα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επομένων μηνών. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, έκανα μια μικρή ανασκόπηση των προτεραιοτήτων της ελληνικής προεδρίας στο επαιδείο των εργασιών του Συμβουλίου σε μια σειρά από θέματα αλλίες τα οποία έχουμε να χειριστούμε τους επόμενους μήνες. Στη συγκυρία των ευρωεκλογών, μια διαδικασία φυσικά ιερή και δηλωτική της δημοκρατίας που διέπει τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί για μας πρόκληση να εργαστούμε με ρεαλισμό και με την πεποίθηση για ένα καλό αποτέλεσμα. Θέλουμε μια αποτελεσματική προεδρία. Βασιζόμαστε για το σκοπό αυτό στη στενή και την ενεργό συνεργασία με το Ευρωκοινοβούλιο που είναι απαραίτητη ώστε να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τους στόχους μας και να μπορέσουμε από κοινού να βρούμε λύσεις σε μια σειρά από σημαντικά και ευαίσθητα θέματα τα οποία θίξατε και εσείς και εγώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Κύριε Πρόεδρε, με πολύ χαρά θα δεχτώ ερωτήσεις που ενδεχόμενα είτε εσείς έχετε είτε έχουν τα μέλη της Επιτροπής σας. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Και τώρα θα ξεκινήσουμε με τον πρώτο γύρο παρεμβάσεων. Επειδή δεν μου ζήτησαν τίποτα οι συντονιστές. Θα ξεκινήσουμε με τη σειρά που ζητούν το λόγο. Η κυρία Πατράο Νέβες καταρχάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, εχθές Σας ευχήθηκα καλή επιτυχία για την Προεδρία σας και το επαναλαμβάνω και σήμερα. Εχθές ήμουν στην Επιτροπή Γεωργίας, σήμερα εδώ. Ε, σας είπα εχθές ότι διάβασα το πρόγραμμα της Ελληνικής Προεδρίας και τις συγκεκριμένες προτάσεις για τη Γεωργία, αλλά διάβασα και τις συγκεκριμένες προτάσεις για την Αλία. Και σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι το πρόγραμμά σας είναι πρόγραμμα το οποίο ε, συμμεριζόμαστε και εμείς και πραγματικά θα θέλαμε να εφαρμοστεί. Δικαίως εσείς μας είπατε ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι και θα θέλατε να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Και συνειδητοποιείτε και πλήρως ότι το συγκεκριμένο εξάμεινο θα είναι μάλλον σύντομο. για να μπορέσει τουλάχιστον να συνεχιστεί η συνεργασία με το Σύνομο συνομοθέτη, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι εμείς θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας μέχρι τις 17 Απριλίου και μετά θα υπάρξει διακοπή για τις ευρωεκλογέ. Ε, συμφωνούμε σε γενικές γραμμές με τα όσα μας είπατε, αλλά όλα αυτά ε, προϋποθέτουν και μια περαιτέρω δέσμευση και από πλευρά σας και από πλευρά μας, διότι θέλουμε και εμείς να ολοκληρώσουμε τη θητεία μας ε, έχοντας επιτύχει τους στόχους που είχαμε προκαθορίσει και πολλοί από αυτούς είναι πολύ σημαντικοί. Παραδείγματος χάρη το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλείας. Δεν ήξερα βέβαια ότι θα λάβω πρώτη το λόγο, διότι είχα την ελπίδα ότι ο κύριος Καντέκ θα ε, μιλούσε πριν από μένα και θα σας έλεγε λίγα περισσότερα ε, για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο εισηγητής βέβαια θα πει περισσότερα. Εγώ να πω απλώς ότι προφανώς αποτελεί προτεραιότητα το θέμα του ταμιολίας. Και γιατί το όλο θέμα της ε, μεταρρύθμισης της κοινής αλληλευτικής πολιτικής ε, είναι άχρηστο εάν δεν εγκριθεί ο κανονισμός για το Ταμείο Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Μας απογοήτευσαν λίγο όλα όσα συνέβησαν στα τέλη του Δεκεμβρίου και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να μπορέσουν να αντιληφθούν ότι όπως προβλέπονται και από τις συνθήκες, ο τριμερής διάλογος θα πρέπει να είναι ακριβώς διάλογος. Ο συνάδελφος Καντέκ μάλλον θα σας πει περισσότερα για το ζήτημα βέβαια. Υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο μας ε, ανακοινώσετε κύριε Υπουργέ και μας ανησυχεί ιδιαίτερα τα πολυετή σχέδια διαχείρισης. Υπάρχει σχετική ε, ψηφοφορία και όπως είπαμε και χθες μας ανησυχεί ιδιαίτερα το θέμα αυτό. Τους τελευταίους μήνες συζητήθηκαν μόνο ε, τα πολιτή σχέδια διαχείρισης ε, για μεμονωμένα είδη, αλλά υπάρχουν πάρα πολύ περισσότερα πράγματα, ε, τα οποία μας πιέζουν πολύ περισσότερα από πλευράς χρονικής. Ελπίζουμε λοιπόν να μπορέσουμε να συνεργαστούμε για να επιληθεί επιτέλους ένα πρόβλημα το οποίο το σέρνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εάν δεν γίνει κάτι, εάν δεν εφαρμοστούν τα πολιετή σχέδια διαχείρισης, ε, δεν θα μπορέσει να ευοδοθεί η κοινή αλληλευτική πολιτική και όλη η μεταρρύθμιση. Και δύο σύντομες παρατηρήσεις τώρα. Οι αλληλευτικές συμφωνίες. Είναι ουσιώδης η εξωτερική διάσταση της αλληλευτικής πολιτικής. Γι' αυτό και εμείς θα πρέπει να ε, παραμείνουμε σταθεροί στις αρχές μας και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση ε, να τις απαρνηθούμε για τις αλληλευτικές συμφωνίες. Οι νέες ε, αλληλευτικές συμφωνίες σε κάποιες περιπτώσεις περιορίζουν τις αλληλευτικές δυνατότητες και αυξάνουν το ε, ποσοστό συγχρηματοδότησης, το ποσοστό της συμμετοχής. Αναφέρομαι και πάλι στο Ταμείο Αλίας. Ε, ο Αλέν ε, ελπίζω να μην με παρεξηγήσει. Πρέπει όμως να το θίξω το θέμα αυτό, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας, κυρίως ποσοστά ανεργίας των νέων και επομένως οποιαδήποτε δυνατότητα μπορεί να τους προσφερθεί. Χάρη στο Ταμείο Αλίας ε, για τους νέους στον τομέα της Αλίας είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτό φυσικά συμβαδίζει και με την κατάλληλη κατάρτιση. Διότι το μεγάλο στίχημα στον συγκεκριμένο τομέα για τους νέους αποτελεί και στίχημα υπέρ της βιωσιμότητας της αλίας. Επομένως, θα πρέπει να προσφέρουμε μια εγγύηση θέσεων εργασία για τους νέους, οι οποίες θα είναι και βιώσιμες. Το να μπορέσουμε λοιπόν να ανανεώσουμε το συγκεκριμένο κλάδο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ για τις προτεραιότητές σας και καλή τύχη. Έχω έξι άτομα που έχουν ζητήσει το λόγο, ο Πρόεδρος. Ε, θα ήθελα να επικεντρωθείτε στις συγκεκριμένε ερωτήσεις που θέλετε να θέσετε στον Υπουργό για να έχει και χρόνο να σας απαντήσει, διότι μέχρι τις 4.30 έχουμε περίπου χρόνο. Ε, τρία λεπτά λοιπόν για τον κάθε μιλητή νομίζω ότι αρκούν. Ο κύριος Στίβενσον και μετά ο κύριος Αρσένης. Ο κύριος Στίβενσον πρώτα. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλωσορίζω και εγώ τον ε, Υπουργό και θα ήθελα ακριβώς να απηχήσω και εγώ αυτά που ίσως ήδη ακούστηκαν σχετικά με τα πολιετή σχέδια διαχείρισης. Εσείς στην εισαγωγή σας κύριε Υπουργέ τονίσατε τη σημασία των πολιετών σχεδίων για να επιτύχει η μεταρρύθμιση της κοινή αλλιευτικής πολιτικής. Γι' αυτό ευχαριστώ την ελληνική προεδρία για τον ενθουσιασμό τον οποίο ε, επέδειξε με στα πλαίσια της Task Force. Εσείς φτάνετε τώρα ε, και αναλαμβάνετε τα ενία στο πιο δύσκολο κομμάτι με, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα διότι όπως είπε και η Μαρία σε τρεις μήνες ε, και σταματούν, οι διακόπτονται οι εργασίες του Κοινοβουλίου. Μέχρι το τέλος Μαρτίου είναι πάρα πολύ δύσκολο να ε, κάνουμε δουλειά. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστώ για τον ενθουσιασμό σας. Είναι ζωτική σημασία πάντως. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτές τις, ε, με, με, με, τις μονομαχίες ε, τύπου Gladiator που είδαμε το Δεκέμβρη στο Συμβούλιο. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστούν αυτά. Ε, δεν μπορούμε πρέπει να αφήσουμε να βοηθήσουμε τους αλληλείς τους ώστε να μπορούν να πάνε κάποια στιγμή στην τράπεζα να πάρουν ε, χρήματα ή κάποιο δάνειο για να ανανεώσουν τα εργαλεία τους αν μη τι άλλο ελπίζω λοιπόν ελπίζω να μπορέσουμε να ε, επιτύχουμε τους στόχους μας επιτυχώς σχετικά με τα πολυετή σχέδια διαχείρισης και ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι στην Ελληνική Προεδρία για τον τρόπο που προσεγγίζει το θέμα. Euh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Είμαι εισηγητή για το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Θάλασσα και Αλία. Έχουμε ακριβώς τους ίδιους στόχους. Εσείς και εμείς. Να καταλήξει δηλαδή το ταχύτερο δυνατό το θέμα αυτό. Φυσικά για να γίνει αυτό πρέπει η Επιτροπή και το Συμβούλιο να κάνουν την αναγκαία προσπάθεια. Υπενθυμίζω ότι είχαμε καταλήξει σε συμφωνία, αλλά δυστυχώς η συμφωνία αυτή τροποποιήθηκε μεταξύ Τυρού και Αχλαδίου για λόγους που δεν γνωρίζω. Και μίλησα στο τηλέφωνο επί μακρόν την προηγούμενη εβδομάδα με την Επίτροπο κυρία Δαμανά και εκείνη μου τηλεφώνησε, ανταλλάξαμε απόψεις και με πληροφόρησε ότι είναι διατεθειμένη να κάνει ό,τι μπορεί ιδιαίτερα για την άμεση διαχείριση που ήταν κάτι που ε, προκαλούσε ε, εμπόδια σε επίπεδο της Κομισιόν. Ε, σημείωσα τις προτάσεις και πριν από λίγο μερικά λεπτά, λεπτά συναντήθηκα με τον Λόρι Evans και την κυρία Χριστοφίδου που είναι η επικεφαλής του ιδιαίτερου γραφείου της κυρίας Δαμανάκη που με επιβεβαίωσαν αυτή την στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει μια δυναμική και από πλευράς Κοινοβουλίου και Επιτροπής για να επιληθεί το θέμα αυτό, να επιτύχουμε κάτι, να πείσουμε το Συμβούλιο, το οποίο εκπροσωπείτε εσείς κύριε Υπουργέ, να συμμετάσχει σε αυτή τη δυναμική για να καταλήξουμε για αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι αν το Συμβούλιο έχει την ίδια αντιμετώπιση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί να μην ξαναρχίσουμε και γιατί να μην καταλήξουμε σύντομα τον τριμερή διάλογο. Αλλά υπενθυμίζω ότι βεβαίως με τη στήριξη και τη συμφωνία όλων των σκιωδών εισηγητών συναδέλφων μου αποφασίσαμε να αναστείλουμε τις διαπραγματεύσεις το Δεκέμβριο. Δεν είναι γιατί μας άρεσε. Είναι, είναι διότι οι προτάσεις που μας είχαν υποβληθεί ήταν απόλυτα απαράδεκτες για το Κοινοβούλιο τις προτάσει του Συμβουλίου και τη Επιτροπή σε εκείνη τη φάση. Υπενθυμίζω ότι είχα τη στήριξη όλων των πολιτικών ομάδων τότε και του Προέδρου του Κοινοβουλίου, του κυρίου Μάρτιν Σούλτ, που με, που με διαβεβαίωσε ότι με στηρίζει. Επαναλαμβάνω και ε, εφόσον έχω αυτή την εντολή ε, που μου ε, εμπιστεύτηκε το Κοινοβούλιο, είμαστε διατεθειμένοι να ξαναρχίσουμε τι διαπραγματεύσει και να καταλήξουμε τάχιστα, γιατί ξέρουμε όλοι ότι είναι απόλυτα αναγκαίο για τι χώρε και για του αλληλεί μας, για τον κλάδο. Αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Θάλασσα και Αλίας να δημιουργηθεί όσο δυνατόν πιο σύντομα. Με βάση λοιπόν ε, το ότι το, η Επιτροπή είπε ότι θα κάνει μια προσπάθεια και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι και το Συμβούλιο θα κάνει προσπάθεια πιστεύω ότι θα πρέπει να ξαναξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Ε, θα γίνει μια άτυπη ανταλλαγή ανταλλαγή αύριο μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής για να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε το πλαίσιο που θα μας επιτρέψει, ελπίζω, την επόμενη εβδομάδα να ξαναξεκινήσει ο τριμερής διάλογος. Ε, αναφερθήκατε στο Μάρτιο, τον Απρίλιο. Εγώ θα επιθυμούσα να καταλήξουμε τον τρέχοντα μήνα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Καντέκο. Ο κύριος Αρσένης. Παρακαλώ. Να σας καλωσορίσω Υπουργέ στην, ε, στο Κοινοβούλιο και στην ε, Επιτροπή Αλληλείας. Ε, το Κοινοβούλιο καλωσορίζει θερμά την Ελληνική Προεδρία και θα είναι στο πλευρό της για να πετύχει τους φιλόδοξους στόχους που έπρεπε και έχει βάλει. Η επιτυχία κάθε Προεδρίας είναι πόσους φακέλους σημαντικούς καταφέρει να κλείσει και πραγματικά βλέπω ότι έχετε βάλει δύο από τους ε, φακέλους που μας απασχόλησαν πάρα πολύ σε αυτή την ε, επιτροπή και το Ταμείο ε, Αλίας που μόλις μίλησε ο κ. Καντέκ αλλά και την αλία βαθέων υδάτων ε, που είχα τη χαρά να είμαι εισηγητής. Και βλέπω ότι έχετε βάλει και τους δύο φακέλους αυτούς σε προτεραιότητα. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια συνταγή επιτυχίας και σας την εύχομαι με όλη μου την καρδιά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Σένη. Κύριε Λεβίν. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τον Υπουργό στην Επιτροπή μας και να ευχαριστήσω για αυτά που είπατε ότι θέλετε δηλαδή να συνεργαστείτε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. πολύ σημαντικό σημαντικός ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, ανα, αναγνωρίζεται και όλα ότι έχουν αυξηθεί οι αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου ε, τώρα για την εξωτερική πτυχή της αλληλευτικής πολιτικής. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική και χαίρομαι που το ίδιο πιστεύετε κι εσείς. Μιλήσατε για τις διαπραγματεύσεις με τη Μαυριτανία και τη Σενεγάλη. Χαίρομαι γι' αυτό και ελπίζω ότι θα ε, βασιστούμε κατά τη διάρκεια της διαπραγματεύσεως στις βασικές αρχές της νέας κοινή αλλιευτικής πολιτικής για... και θα επιμείνουμε στην πλεονασματική ποσότητα ε, ηχθείων που δεν χρειάζεται για εσωτερική κατανάλωση η χώρα κτλ. Για να μπορέσουμε να έχουμε βιώσιμη αλία παντού. Αναφερθήκατε στους διάφορους κανονισμούς ε, και εγώ ήμουνα ε, εισηγήτρια για το σχέδιο ανάκαμψης του αποθέματος των χελιών. Ε, βέβαια δυστυχώς από τότε που ε, εγκρίθηκε ο, ε, εγκρίθηκαν τα σχετικά στη, πέρσι στην Ολομέλεια δεν έγιναν και πολλά πράγματα. Το άλλο θέμα είναι η χρηματοδοτική πτυχή, πράγματι διατίθεται κονδύλια από το Ταμείο για τους ελέγχους, και υπάρχει και προβλέπονται και κάποια κονδύλια φαντάζομαι για την άμεση διαχείριση ε, κατά, υπά, προτείνεται μια κατανομή των κονδυλίων αλλά δεν ξέρω εσείς ως υπουργός τι πιστεύετε. Πιστεύετε περισσότερα κονδύλια προέρθουν από την άμεση διαχείριση ή από πού, τι πιστεύετε γι' αυτά. Τώρα, αναφερθήκατε στον κανονισμό Omnibus που λέμε και στην απαγόρευση των απορρίψεων. Το Συμβούλιο θα καταφέρει να πάρει τελική θέση ε, στο εξάμεινο της Προεδρίας σας θα φαντάζομαι ότι αυτό θα είναι δύσκολο βέβαια λόγω των ευρωεκλογών αλλά για το Omnibus ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της ελληνικής προεδρίας και τώρα για το IMP και τα λοιπά είναι καλό που δίνει προτεραιότητα στο θέμα η προεδρία εσείς θα προχωρήσετε με την ε, οδηγία για το χωροταξικό σχεδιασμό. Να καλωσορίσω πριν δώσω το λόγο στον επόμενο μιλητή σε μια ομάδα ε, φοιτητών, ε, φοιτητών πολιτικών επιστημών που είναι εδώ, προσκεκλημένη της κυρίας Τόμα. Ε, σας καλωσορίσουμε λοιπόν και είναι εξαιρετική ευκαιρία που είστε εδώ μαζί με τον Υπουργό. Κύριε Τομάν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ με τη σειρά μου να καλωσορίσω τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου και να του πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω ότι το πρόγραμμά του είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο, διότι αν δεν κάνω λάθος, ε, τρεις μήνες και κάτι έχει στη διάθεσή του για να το ολοκληρώσει με τη βοήθειά μας και Χαίρομαι διότι οι προτεραιότητες που ανακοινώσατε είναι πολύ συμβατές με το χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής μας. Και εδώ να συμφωνήσω με αυτό που είπε και η κυρία Πατράου. Σίγουρα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας αποτελεί προτεραιότητα. Νομίζω ότι είναι η βασική προτεραιότητα για δύο λόγους. Πρώτον, διότι είναι απαράδεκτο ε, να ε, θεωρήσουν ε, ότι οι πολίτες μας ότι επειδή έχουμε μικροκαυγαδάκια διακυβεύεται το μέλλον ε, της αλίας και το οικονομικό μέλλον της αλίας και οι πολίτες μπορεί να θεωρήσουν ότι όντως αυτοί είναι απλοί, μικρές, απλές διαμάχες. Και επίσης αν δεν καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία πολύ σύντομα μέχρι το τέλος της θητείας θα ξεκινήσει η διαδικασία εκ του μηδενός και αυτό και πάλι θα είναι εις βάρος των πολιτών. Χαίρομαι λοιπόν που θα ασχοληθείτε και ε, με τον κανονισμό ε, για την αλία βαθών υδάτων και με ενδιαφέρει και το θέμα της Νορβηγίας. Όπως είπατε κι εσείς, ε, οι συμφωνίες με την Νορβηγία είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για όλη την αλία του Ατλαντικού. Έχουν συνέπειες και στην κοινή πολιτική και στα τάκ και στις ποσοστώσεις και φυσικά οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι τελείως κρυφές. Ε, ξέρω ότι δεν υπάρχει νημοκή υποχρέωση, δεν προβλέπεται καν το Κοινοβούλιο να λαμβάνει γνώση του τι συμβαίνει ε, σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, αλλά επειδή υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές συνέπειες οι οποίες ε, θα προκύψουν από αυτές τις συμφωνίες για την αλία μας, θα έπρεπε ίσως να έχουμε κάποιες περαιτέρω διευκρινήσεις, κάποια περισσότερη διαφάνεια για το μέλλον αυτών των διαπραγματεύσεων και το πώς προχωρούν. Ευχαριστώ η κυρία Ρόντουστ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Από πλευρά της ε, πολιτικής ομάδα, ομάδας, της ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών σας καλωσορίζω και χαίρομαι πολύ που έχετε αναλάβει την Προεδρία. Βλέπω ότι ε, φιλόδοξους ε, στόχους έχετε θέσει, πολλά υπόθηκαν. Θα πω λοιπόν και εγώ συνοπτικά η ομάδα μου θεωρεί επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό να διαμορφωθεί έτσι η συμφωνία για την αλληλεία, ούτως ώστε να διαμορφώνονται έτσι οι συμφωνίες για την αλληλεία, ούτως ώστε να μην αφαιρούμε τα μέσα διαβίωσης από άλλους αλληλείς. Αλλά θα έπρεπε να επιτρέπουν αυτές οι συμφωνίες αλληλείας να μην φεύγουν από τις χώρες τους ε, κάποιοι αλληλείς και θα πρέπει ως Κοινοβούλιο και Συμβούλιο να αντιμετωπίσουμε σοβαρά αυτή την εξωτερική διάσταση, γιατί μόνο έτσι θα είναι δυνατόν να μην μεταναστεύουν από τις χώρες τους οι αλληλείς άλλων χωρών. Θα ήθελα να μου πείτε τι προβλήματα βλέπετε να υπάρχουν ακόμη για το Ταμείο. Είπατε πολλά γενικά το Ταμείο για τη θάλασσα και την αλία, αλλά παρακαλώ πέστε μου με τρία-τέσσερα λόγια. Πού βλέπετε να είναι τα κυριότερα προβλήματα για να καταλήξει το θέμα αυτό. Παρακαλώ, επιγόντως, Δεν ήμουν παρούσα χθε στη συνεδρία τη ομάδα εργασία Tax Force, αλλά άκουσα τι συζητήθηκε και με χαρά άκουσα ότι αναλάβατε την δέσμευση να λήξουν οι εργασίες μέχρι τον Μάρτιο. Δεν είμαι απεσιόδοξη από τη φύση μου, αλλά επειδή έχω κάνει πέντε χρόνια στο Κοινοβούλιο, δεν είμαι πια και τόσο αισιόδοξη που να πιστεύω ότι αυτό είναι εφικτό, αλλά θα σας υποστηρίξω. Ξέρετε ότι συζητήσαμε τι θα συμβεί αν δεν υπάρξει συμφωνία με το Συμβούλιο, ότι θα ήμασταν διατεθειμένοι να ε, προσφύγουμε στο δικαστήριο. Δεν μου αρέσει βέβαια αυτό να προσφεύγει μια, ο ένας θεσμός κατά του άλλου, αλλά πρέπει να έχετε υπόψη ότι θα ήμασταν διατεθειμένοι εάν δεν καταλήξουμε σε σόφρονα συμφωνία συντόμως. Τώρα, κανονισμός όμνιμπους. Το συζητάμε πολύ αυτή τη στιγμή και είμαστε ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι με την κατάσταση. Από 1η Πρώτου 15 θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει η απαγόρευση απορρίψεων. Οπότε έχουμε μόνο τρεις μήνες, για, όπως ξέρετε, για να ε, καταλήξει τις εργασίες του αυτό το Κοινοβούλιο και με βάση τον εσωτερικό μας κανονισμό και το άρθρο 2.14 συγκεκριμένα, όλες οι εκθέσεις που δεν έχουν αποφασιστεί, ακόμη και αν συζητώνται, καταπίπτουν όταν λήξει η θητεία. Εκτός εάν η διάσκεψη των Προέδρων πει εκπεφρασμένα ότι κάποιο θέμα μπορεί να εξακολουθήσει να συζητείται. Είναι ιδιαίτερα λυπηρή αυτή η κατάσταση. Και εμείς, αλλά και εσείς, δεν θα θέλαμε να αναλάβουμε την ευθύνη την 1η Πρώτου 15 να απαιτούμε να απαγορευτούν ή απορρίψεις χωρίς να υπάρχει κατάλληλη νομική βάση. Θα μπορούσατε λοιπόν εσείς ε, ως Συμβούλιο να αντιμετωπίσετε το ενδεχόμενο να εγκρίνετε την πρόταση της Κομισιόν υπό την επιφύλαξη ότι θα ισχύσει μόνο για ένα χρόνο, ούτω ώστε το, ένα, το νέο Κοινοβούλιο να έχει επαρκή χρόνο για να καταλήξει σε μια καλή συμφωνία. Αυτά καταρχάς για το σκουμπρί νομίζω ήδη τέθηκε από την κυρία Τομά και για το θέμα αυτό και εγώ θα ήθελα μια συγκεκριμένη απάντηση από σας. Ευχαριστώ. Και, α, ε, Μιλάνα και Γκάλαχερ, παρακαλώ. Μιλάνα, Γκάλαχερ και κλείνουμε και μετά θα δώσουμε το λόγο στον Υπουργό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς όρισατε κύριε Υπουργέ ένας τρόπος και μόνον υπάρχει για να ολοκληρωθεί ο τριμερής διάλογος για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου και εμείς είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε. Έχουμε αποδείξει ε, στη διάρκεια των προηγούμενων τριμερών διαλόγων ότι έχουμε τη δυνατότητα της διαμεσολάβησης, η οποία όμως δεν ε, ήταν αρκετή για τις διαπραγματευτές του Συμβουλίου μέχρι τούδε πάντα είχαν πολύ αυστηρές εντολές και ορισμένες φορές υπήρχαν ε, ε, προσκόμματα τα οποία δεν μπορούσαν να υπερκεραστούν. Εμείς θέλουμε δύο πράγματα ουσιαστικά. Πρώτον, να μην υποβληθεί το Κοινοβούλιο στην ανάγκη να πρέπει να διαβουλεύεται μεταξύ, ε, στο, όσα διαβουλεύονται οι χώρες μεταξύ τους και επίσης Υπάρχει η μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής, την οποία εγκρίναμε και συμφωνήσαμε με το Συμβούλιο. Και υπάρχουν κάποιες ε, ε, στάσεις του Συμβουλίου ε, όταν έρχεται στις διαπραγματεύσεις που θέλουν να διακυβεύσουν αυτά τα δύο πράγματα. Και το μόνο που δεν θέλει να κάνει το Κοινοβούλιο είναι να προδώσει όσα έχει ήδη ε, συμφωνήσει με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο να κλείσουμε πολύ καλά αυτή τη συμφωνία και θα ήθελα να σας δώσω μια συμβουλή αν μου επιτρέπετε. Δεν συνηθίζεται βέβαια να δίνετε συμβουλή σε έναν Υπουργό από το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να έχετε μία εντολή λίγο μεγαλύτερη και να μην είναι τόσο αυστηρή η εντολή σας από πλευρά Συμβουλίου. Διότι αν είναι λίγο περισσότερο, μεγαλύτερο το περιθώριο ευελιξίας, εγώ είμαι πεπισμένος ότι ένας μεσογειακός υπουργό θα μπορέσει να διαμεσολαβήσει ως Μεσόγειος και να καταφέρει να κλείσει ειρηνικά αυτή την υπόθεση. Άλλα δύο θέματα θα ήθελα να σας θέσω. Ζείτε όπως και εγώ στη Μεσόγειο και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει ο κανονισμός για τη Μεσόγειο που τα τελευταία χρόνια έχει καθορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το τι συμβαίνει στη συγκεκριμένη θάλασσα. Ο κανονισμός αυτός ε, σε μεγάλο βαθμό δεν έχει εφαρμοστεί, διότι ίσως κάποια πράγματα δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν. Έχουν περάσει τρία χρόνια από τότε που τέθηκε σε ισχύ. Προβλέπεται ότι θα γίνει μια ε, επαλήθευση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία της αξιολόγησης και επαλήθευσης και ελπίζω στους επόμενες μήνες να έχουμε μια κάποια πρωτοβουλία για την αναθεώρηση του κανονισμού για τη Μεσόγειο. Διότι υπάρχουν δύο αντιφάσεις αυτή τη στιγμή. Αφενός υπάρχει ένας κανονισμός ο οποίος δεν εφαρμόζεται και υπάρχει ένας, ε, ε, ένα καθεστώς ελέγχων ο οποίος πολλές φορές ποινικοποιεί απλώς και μόνον και ε, αφετέρου έτσι όπως είναι διαμορφωμένος αυτός ο κανονισμός ελοχεύει ο κίνδυνος να μην επιτύχει καν η μεταρρύθμιση που έχουμε γκρίνει διότι είναι πάρα πολύ αυστηρά τα πράγματα. Εγώ δεν σας λέω ότι έχω τη λύση σήμερα, απλώς σας λέω ότι ο κανονισμός αυτός έτσι όπως είναι διαμορφωμένος, ο οποίος διαμορφώθηκε και χωρίς συζήτηση με το Κοινοβούλιο, να σας υπενθυμίσω ότι έγινε πριν από τη συνθήκη της Λισαβόνας και τον ε, παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον συζήτησαν απλώς τα κράτη-μέλη χωρίς να συμμετέχει καθόλου το Κοινοβούλιο. Και πρέπει να σας πω, ε, επιτρέψτε μου κιόλας να το πω, ότι το γεγονός ότι δεν υπήρχε το άγρυπνο μάτι του Κοινοβουλίου έχει οδηγήσει σε αυτή τη μορφή του κανονισμού και ελπίζω τους επόμενους μήνες ε, να ε, μιλήσετε κι εσείς με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να αντιμετωπίσετε ανοιχτά αυτή την πιθανή αναθεώρηση. Κάτι τελευταίο. Πριν από κάποιες εβδομάδες ε, εγκρίναμε μία έκθεση για την αλλιευτική στρατηγική στην Αδυρατική θάλασσα και στο Ιόνιο Πέλογος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε ώστε η συγκεκριμένη έκθεση πρωτοβουλία, της οποίας ήμουν εισηγητής και υπερψήφισε το Κοινοβούλιο, ε, δεσμεύτηκε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρουσιάσει μία ε, πρόταση μέχρι τον Ιούνιο. Εμείς περιμένουμε λοιπόν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα κι εσεί ε, να ε, προσέξετε γιατί θέλουμε να έχουμε αυτή την πρόταση, διότι να υπάρχει μια πολιτική για την Αδριατική και το Ιόνιο Πέλαγος είναι πολύ σημαντικό. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δεσμεύεται για την ε, μακροπεριφερειακή στρατηγική Αδριατική Ιωνίου και επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό μαζί και με τα όσα γίνονται για τη Βαλτική. Σας εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία και ελπίζω να ολοκληρωθεί αυτό το εξάμεινο και να μπορέσω να σας δώσω συγχαρητήρια διότι ε, φέρατε σε αίσιο πέρα σε όλες τις πρωτοβουλίες που μας επισημάνατε. Ευχαριστώ ο κύριος Γκάλαγκερ για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Uh, uh, το μικρόφωνο παρακαλούμε. Το μικρόφωνο παρακαλούμε. Ευχαριστώ. Θέλουμε ε, να ευχηθούμε κάθε επιτυχία κατά τη διάρκεια της Προεδρίας που όπως είπατε και εσείς βασίζεται στην ανάπτυξη, την απασχόληση και τη συνοχή. Ο κύριος Υπουργός ε, με συγκίνησε όταν αναφέρθηκε στην σημασία της θάλασσας και της αλίας για τις παράκτιες περιοχές και τα νησιά, όπου υπάρχουν πολύ λίγες δυνατότητες απασχόλησης, άλλες δυνατότητες απασχόλησης και με εντυπωσίασε αυτό που είπε. Αλλά φυσικά θα σας κρίνουμε στο τέλος της θητείας σας, αλλά παρουσιάσατε με μεγάλη διάβια τις προτεραιότητές σας και χαίρομαι γι' αυτό. Τώρα σε σχέση με το Ταμείο Θαλασσιαλίας για να επιμείνω, δεν θέλω να επιμείνω ιδιαίτερα βέβαια, αλλά πρέπει να βρούμε μια λύση. Και υπάρχουν πολλοί που θέλουν να υπάρξει πρόοδος, γιατί αν δεν υπάρξει συμφωνία οι επιπτώσεις είναι, θα ήταν τόσο απέσει που ούτε να τις σκεφτώ δεν μπορώ. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει τριμερής διάλογος. Και τριμερής διάλογος σημαίνει όλοι να έχουν καλή θέληση. Τώρα για τα πολυετή ε, σχέδια διαχείριση είμαι μέλος της ομάδας εργασίας αυτής, Task Force, και είμαι υπεύθυνο για το σκουμπρί της, ε, του βορειοανατολικού Ατλαντικού. Ε, θα ήταν ξεφτύλα να μην καταφέρουμε να κλείσουμε το θέμα αυτό. Και με εντυπωσίασε η στάση των εκπροσώπων σα στη μόνιμη αντιπροσωπή όταν του είδαμε χθε. Και φυσικά αν δεν επιτύχει η προσπάθεια αυτή δεν θα φταίνει εκείνη. Αλλά όπω με όλα τα πράγματα στη ζωή πρέπει να αντιμετωπίσουμε πρώτα τα απλούστερα. Το απλούστερο ήταν ε, ένα μόνο είδο, μετά ήταν δύο είδη. Τώρα όταν περνάμε στη μεικτή αλληλεία είναι πολύ πιο περίπλοκο, αλλά με εντυπωσιάζουν προσπάθειες και των τριών θεσμικών οργάνων για να κλείσει το θέμα αυτό μέχρι τέλη Μαρτίου υπό την προεδρία σας και υπό την προεδρία του Stuart Στίβενσον. Τώρα για τον ε, κανονισμό Omnibus. Φυσικά όλοι θέλουμε να συνεργαστούμε, αλλά μπορούμε να καταλήξουμε μόνο εάν εργαζόμεθα νομοτύπως. Ίσως λοιπόν να μην μπορέσει να ξεκινήσει η εξέταση του θέματος αυτού παρά μόνο μετά τις εκλογές. Γιατί όπως ξέρετε ό,τι συζητάμε τώρα ε, καταπίπτει όταν κλείσει η θητεία. Ένα μεγάλο θέμα για μας ε, εδώ και αρκετά χρόνια είναι η βιωσιμότητα διαφόρων ε, και, και εγώ και άλλοι συναδελφοί μου ανησυχούμε πολύ για τη βιωσιμότητα του σκουμπριού στον βορειοανατολικό Ατλαντικό. Ξέρω ότι σήμερα συναντώνται στο Λονδίνο οι χώρες της περιοχής και δεν ξέρω μήπως έχετε καμία ενημέρωση. Ε, αν δεν έχετε το καταλαβαίνω, αλλά θα θέλαμε να μάθουμε τι γίνεται τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Γκάλαχερ. Κύριε Υπουργέ, ήταν πολλές οι ερωτήσεις. Ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Ε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό δείχνει και το ενδιαφέρον και την ποικιλία των θεμάτων που έχουμε να συζητήσουμε για τα θέματα της αλίας. Ε, θα μου επιτρέψετε μόνο να καλωσορίσω και εγώ τους φοιτητές. Προφανώς οι φοιτητές έμαθαν ότι ο νέος Υπουργό για τη Γεωργία και την Αλληλεία της στο Συμβούλιο είναι καθηγητής και ήρθαν για υποστήριξη του καθηγητή της. Τώρα έρχομαι κατευθείαν στο πιο σημαντικό θέμα που θίξατε όλοι και είναι αυτό ε, με, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Θάλασσα και την Αλία. Ειλικρινά σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας, γιατί όλα τα σχόλια και ακόμα και οι ερωτήσεις που τέθηκαν, τέθηκαν με έναν επικοδομητικό τρόπο να βρούμε μία λύση και να ολοκληρώσουμε αυτή τη συμφωνία. Είμαστε απόλυτα δεσμευμένοι με την, για τη συνέχιση αυτών των διαπραγματεύσεων με το Κοινοβούλιο και με την έβρεση συμβιβαστικής λύσης, ε, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία. Είμαι στεπεπισμένη ότι όλοι μας μοιραζόμαστε την ίδια επιθυμία. Το άκουσατε εσείς από μένα, το άκουσα εγώ από εσά και μπορώ να διαβεβαιώσω όπως έκανε και ο κύριος Καντέκ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυρία Δαμανάκη είναι της ίδιας άποψης. Πρέπει ο τρίλογος να καταλήξει κάπου για να κλείσει αυτή η συμφωνία. Γιατί μη έχοντας τη συμφωνία δεν έχουμε ταμείο και χωρίς ταμείο δεν έχουμε αλλιευτική πολιτική αυτή την ώρα. Επομένως πρέπει γρήγορα να κλείσει αυτό το θέμα. Και είμαι σίγουρος ότι θα διαργαστούμε και με διαφάνεια και αποκλειστικό στόχο να βρεθεί μια ικανοποιητική λύση για όλους και όπως πληροφορήθηκα ήδη έχει προγραμματιστεί μια πρώτη συνάντηση αύριο πέμπτη, σας το ανέφερα ήδη, άρα δείχνει ότι βιαζόμαστε και θέλουμε να κλείσουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε. Για όλα τα κρεμή ζητήματα των διαπραγματεύσεων για το Ταμείο, όπως προανέφερα, οι απόψεις των θεσμικών οργάνων και φυσικά και του Κοινοβουλίου θα αποτελέσουν την ουσία της συζήτησης και από κοινού θα δογηθούμε στη λύση. Πάντως θέλω να πω ότι εγώ τουλάχιστον σας δηλώνω ότι επιδιώκουμε αυτή την πολιτική συμφωνία μέχρι το τέλος του μήνα δείχνοντας έτσι την ισχυρή δέσμευσή μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας. Μην ξεχνάτε ότι επειδή θύχθηκε και το θέμα της ανεργίας, των νέων κλπ. Πολλά πράγματα από αυτά που συζητάμε θα ε, εξαρτώνται από αυτή τη συμφωνία. Ναι, το Ταμείο πρέπει να υποστηρίξει τους νέους. Το κάναμε και για την κοινή αγροτική πολιτική, όπου έχουμε συμφωνήσει βλέποντας τη δημογραφική γύρανση των ανθρώπων που ασχολούνται με το πρωτογενή τομέα, πόσο ανάγκη έχει υποστήριξης νέων ανθρώπων να μπουν στον παραγωγικό ιστό της Ευρώπης, γι' αυτό και αποφασίσαμε και εκεί τουλάχιστον έστω έως 2% των χρημάτων να δοθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το, το θέμα των, ε, των, ε, της αλληλείας των βαθαίων υδάτων που έθιξε και ο κύριος ε, Αρσένης, μη σας εκπλήσει, το κάναμε παρά το ότι γνωρίζαμε τη δυσκολία γιατί πιστεύουμε ότι οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την έναρξη αυτών των εργασιών του Συμβουλίου σε τεχνικό επίπεδο και ήδη λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες που ψήφισε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύουμε ότι παρά το ότι καθυστέρησε, καθυστερεί κάποιος να καταπιαστεί με αυτό το θέμα εδώ και δύο χρόνια, είναι καιρός και έχει φτάσει η οριμότητα να καταπιαστούμε με την αλία των βαθαίων υδάτων και να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε και για αυτό το δύσκολο θέμα. Γι' αυτό το φέραμε και στην προτε... τις προτεραιότητες της Προεδρίας μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα, θέματα των πολιετών σχεδίων διαχείρισης που θίξατε, Δεδομένων των χρονικών περιορισμών που έχουμε λόγω της διακοπής των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ελληνική Προεδρία προτίθεται να συνεχίσει τις εργασίες μέχρι και το τέλος Μαρτίου. Επίσης, έχουμε προγραμματίσει να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της Task Force στου υπουργού του Συμβουλίου Υπουργών του, το Απριλίου. Έτσι, ευελπιστούμε θα προχωρήσουμε και στα πιο πολύπλοκα σχέδια διαχείρισης και να καλύψουμε και τους μικτούς τύπους. Εγώ συμφωνώ και αυτή είναι και η δικιά μου πρόθεση. Έτσι είναι και ο σωστός τρόπος να κινηθούμε. Δεν προσπαθούμε να επιλύσουμε ένα πολύπλοκο πρόβλημα προσπαθώντας να το λύσουμε στην πιο πολύπλοκη του μορφή. Ας μάθουμε, ας το πούμε πιλωτικά και αποκτώντας εμπειρία να το λύσουμε στα απλούστερα θέματα και με την εμπειρία αυτή να πάμε σε ακόμα πολυπλοκότερες καταστάσεις. Πάντως θέλω να τονίσω και σε εσά αυτή είναι και η, απόφασή μας, ότι είμαστε προσιλωμένοι σε αυτό το στόχο. Θέλουμε να βρεθεί λύση στο δια, διαθεσμικό αυτό αδιέξοδο και να συνεχίσουμε την παράδοση μιας ε, πιο καλής θέλησης από όλα τα μέρη προκειμένου να προωθηθούν τα σχέδια αυτά διαχείρισης όπως είπα που είναι πολύ σημαντικά γιατί είναι σημαντικά και για την ανασύσταση των αποθεμάτων και γιατί, που είναι συνειφασμένα με την βιωσιμότητα της αλληλείας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα των ε, απορρίψεων που θύχτηκε από αρκετούς, θέλω να πω ότι όπως ανέφερα, η εξέταση της πρότασης του κανονισμού έχει ήδη ξεκινήσει στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου και πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος της Προεδρίας μας θα ολοκληρώσουμε την εξέτασή της. Θα θέλαμε επίσης να τονίσουμε ότι είναι σημαντικό να έχουμε τον κανονισμό στο τέλος του χρόνου, διότι η υποχρέωση τίθεται σε εφαρμογή, όπως γνωρίζουμε όλοι, από την 1η Ιανουαρίου του 2015. Άρα θα πρέπει να προχωρήσουν οι εργασίες και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το σκοπό αυτό. Ιδιαίτερα τώρα για τον κανονισμό της ε, Μεσογείου που θύχτηκε από τον κύριο Μιλάνα για την αναθεώρηση του κανονισμού για τη Μεσόγειο είναι μια ερώτηση για την Επιτροπή. Άρα ουσιαστικά είμαστε σίγουροι ότι θα μπορέσει να μας απαντήσει για αυτό το θέμα και εμείς θα εργαστούμε μαζί σας προς την κατεύθυνση αυτή προκειμένου να προχωρήσουμε εις ό,τι αφορά και τον κανονισμό αυτό για την Μεσόγειο. Για τις αλληλευτικές συμφωνίες, όπως είπα, θα στηριχτούμε στις αρχές που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της νέας κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Σας διαβεβαιώνω όμως ότι θα έχετε πάντα πλήρη ενημέρωση προκειμένου το Κοινοβούλιο να παρακολουθεί από κοντά αυτές τις εξελίξεις και φυσικά να συμβάλλει και με τη γνώση του και την εμπειρία και φυσικά να εκφράσει και τις απόψεις του για το θέμα αυτό για τα χέλια που θίξατε θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να προχωρήσουμε τις εργασίες και σε αυτό το φάκελο. Ανέφερα προηγουμένως πώς ξεκινήσαμε και ανέφερα ότι μας ενδιαφέρει να προχωρήσουμε γρήγορα και σε άλλους τέτοιους ε, ε, φακέλους. Τώρα τελειώνοντας γιατί έχουμε δύο ακόμα θέματα που αφορούν το, το Σκουμπρί και το Βόρειο ε, Ατλαντικό. Γνωρίζω ότι οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Ως Προεδρία ευελπιστούμε να βρεθεί σύντομα λύση για το θέμα και πιστεύω ότι να είναι ικανοποιητική αυτή η λύση και για, για όλες τις πλευρές. Πάντως είναι ένα σημαντικό θέμα και τελειώνω κύριε Πρόεδρε και ζητώ συγγνώμη που αν παίρνω ένα λεπτό παραπάνω σε ό,τι αφορά το θέμα της ε, Αδριατικής και του Ιωνίου μας ενδιαφέρει και μας και σαν χώρα είναι πράγματι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία και μπορεί να αποτελεί και μια από τις κύριες προτεραιότητες αποτελεί σίγουρα μια από τις κύριες προ, προτεραιότητες και μπορεί να είναι και μια συμφωνία πρότυπο που μπορεί να βοηθήσει και σε παρόμοιες άλλες καταστάσεις. Δεν θέλω να σας πάρω πολύ περισσότερο χρόνο. Σας ευχαριστώ ειλικρινά για, την, για τον χρόνο σας και σας ευχαριστώ για τη βοήθεια εκ των προτέρων κύριε Πρόεδρε και εσάς και τα μέλη της Επιτροπής σας. Ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Πρόκειται για μια εξαιρετική συνάντηση και ανταλλαγή απόψεων και όπως ε, πολύ σωστά είπατε, συμφωνώ και εγώ, ελπίζω στους επόμενες μήνες, στο ε, χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, εδώ ε, με την Επιτροπή μας να μπορέσουμε να έχουμε μια στενή σχέση και συνεργασία. Ευχαριστούμε πολύ και καλή επάνωδο στη χώρα σας. Thank you.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 Συνεχίζουμε λοιπόν με την ημερήσια διάταξη. Λίγο ησυχία παρακαλώ. Να περάσουμε στο σημείο 2. Όπως σας είπα θα ξαναδούμε τα σημεία αυτά. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Η αρχική εκδοχή που λάβατε είχε κάποια ζητήματα. Καταρχάς να σας πω ότι στην αρχή των ψηφοφοριών θα υποβάλουμε και προσψήφιση το σχέδιο ψηφίσματος ε, για την ε, περίπτωση ε, του σκουμπριού στην Βόρεια Θάλασσα είχαμε προβλέψει να πάει για την επόμενη Ολομέλεια και δεν το είχαμε εγκρίνει εδώ στην Επιτροπή μας, επομένως πρέπει να ψηφίσουμε και το θέμα αυτό. Και επίσης υπάρχει και κάτι ακόμα, το 14 και το 15 θα τα ανταλλάξουμε. Θα συζητήσουμε πρώτα το σημείο 15 της κυρίας Μαρία ε, Πατραονέβες ε, για το πρωτόκολλο και τον καθαρισμό των ελευτικών δυνατοτήτων και μετά το 14 της κυρίας Τομάς ε, για τη σύμβαση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Θα ανταλλάξουμε απλώς τα δύο σημεία. Και τέλος, για τις αλληλευτικές ε, προοπτικές ε, στην Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ταϊλάνδης, που είμαι εισηγητής εγώ, ζήτησα να αναβληθεί για τους εξής λόγους. Καταρχάς ε, θεωρώ ότι συμφωνούμε στο μεγαλύτερο τμήμα της έκθεσης. Ε, είχα κάποιες συναντήσεις με κάποιους και αλλά υπάρχουν μια σειρά από αποχρώσεις τις οποίες θα ήθελα να ε, συζητήσουμε για να έχουμε στο το δυνατόν μεγαλύτερη συνένεση. Επειδή λοιπόν έχουμε λίγο χρόνο, ε, θα ήθελα να το αναβάλουμε μέχρι την επόμενη συνεδρία της Επιτροπή μας και την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε κάποιες συναντήσεις με τους κοιόδης ώστε να μπορέσουμε να κλείσουμε ε, το θέμα αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπίσουμε και ιδιαίτερε δυσκολίες. Η κυρία Φράγα, στην ημερήσια διάταξη ζητάμε έτσι. Θα ήθελα να δω αν μπορούμε να συμπεριλάβουμε και ένα σημείο στο τέλος για την ε, Task Force ε, για να μας ενημερώσει για το πώς πηγαίνουν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Θα ήθελα να ενημερωθούμε, διότι δεν γνωρίζω πολύ καλά πώς ε, προχωρά το θέμα και θα ήθελα να το συζητήσουμε. Δεν ξέρω αν ο κύριος Στίβενσον μπορεί αύριο ή όποτε μπορεί να μας ενημερώσει για το ζήτημα. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Στίβενσον. Είχαμε προβλέψει ούτως ή άλλως σήμερα στη συνεδρίαση των συντονιστών την οποία θα συνεχίσουμε μετά την ψηφοφορία. Ε, θα υπάρξει μια ενημέρωση για να δούμε πώς πάει το πράγμα και από εκεί και πέρα εγώ από πλευρά μου δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ε, νομίζω ότι θα έχουμε χρόνο. Ε, η ημερήσια διάταξη μας επιτρέπει να συζητήσουμε και το θέμα αυτό και αν συμφωνεί και ο κύριος Στίβενσον και από ό,τι βλέπω γνέφει καταφατικά ε, θα βρούμε κάποια στιγμή, θα το συμπεριλάβουμε και αυτό στην ημερήσια διάταξη, θα γίνει ενημέρωση ή και στα διάφορα δεν χρειάζεται καν να βάλουμε ξεχωριστό σημείο στην ημερήσια διάταξη. Θα εξαρτηθεί από τον κύριο ε, Στίβενσον, αν θα είναι εδώ για να μας ε, ενημερώσει. Δεν υπάρχει πρόβλημα από πλευρά του κυρίου Στίβενσον, επομένως θα μπορούσαμε να το συμπεριλάβουμε, ίσως να το έχουμε τελευταίο αύριο μετά από την ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Δαμανάκη και την παρουσίαση της έκθεσης. Αύριο λοιπόν θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Για να δούμε στην ημερησία διάταξη. Αύριο το πρωί, στο τελευταίο σημείο του πρωινού, νομίζω ότι θα έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας. Να προσθέσουμε ένα σημείο 16α για να γίνει και ενημέρωση. Συμφωνείτε? Ο κύριος Στίβενσον συμφωνεί. Ωραία λοιπόν, θα προσθέσουμε ένα σημείο 16α, ενημέρωση του κυρίου Στίβενσον για την Task Force. Ωραία. Το εγκρίνουμε και αυτό. Και θα συνεχίσουμε λοιπόν με την ημερήσια διάταξη όπως συμφωνήσαμε. Τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδριάσεων ε, τα έχουμε. Αν δεν υπάρξει κάποια αντίρρηση μέχρι το πέρας της συνεδρίασης, θα θεωρούμε ότι εγκρίνονται. Ανακοινώσεις του Προέδρου να σας πω το εξή. Αύριο το πρωί έχουμε την ψηφοφορία για την έκθεση για την... Ε, ε ειδικέ δράσει τη κοινή ελευθερική πολιτική για την ανάπτυξη του ρόλου των γυναικών. Ξέρετε ότι αυτό το έχουμε από με την Επιτροπή Γυναικών και για να μπορέσουμε να κάνουμε και τη συζήτηση είπαμε να γίνει ψηφοφορία αύριο το πρωί. Αλλά, αυτό είναι το ουσιαστικό, η ψηφοφορία θα γίνει στο 3G3. Θα ψηφίσουμε στην αίθουσα 3G3 και μετά θα επιστρέψουμε εδώ για να συνεχίσουμε με τις συνεδρίες τη Επιτροπή. Έπρεπε να ψηφίσουμε σε μία από τι δύο αίθουσε γιατί είναι κοινή η ψηφοφορία με την Επιτροπή Γυναικών και την Επιτροπή Αλία. Επομένω, κάπου πρέπει να ψηφίσουμε. Θα ψηφίσουμε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση στην αίθουσα στην οποία συνεδριάζει η Επιτροπή Γυναικών την 3G3. Θα ψηφίσουμε στις 9 και μόλις τελειώσει η ψηφοφορία θα επιστρέψουμε εδώ για να συνεχίσουμε με την υπόλοιπη μερίσια διάταξη. Συμφωνείτε, δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση. Ωραία. Περνάμε τώρα στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Ξεκινούμε λοιπόν με τις ψηφοφορίες. Έχετε όλοι τις κάρτες σας. Να ακολουθήσουμε το σύστημα με τις κάρτες, διότι νομίζω ότι είναι καλύτερο από οποιοδήποτε άλλο. Κύριε Γκάλαχερ, δεν έχετε κάρτα μαζί σας. Ωραία. Θα σα ε, προσμετρούμε, να σηκώνετε το χεράκι σα και θα μετρούμε και την ψήφο σα. Κάποια άλλη αντίρρηση. Ωραία. Ξεκινάμε με το σημείο 6 λοιπόν. Vamos a ver. El punto 6 es el que tenemos Σημείο 6. Το σκουμπρί. Α, συγγνώμη. Η πρόταση ψηφίσματος είναι αυτή που δεν είχαμε εδώ. Ε, όπως την είχαμε συμφωνήσει, η πρόταση ψηφίσματος για το σκουμπρί, ε, για την επόμενη ολομέλεια. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε ψηφοφορίας. Εγκρίνεται λοιπόν. Ε, να επαναλάβουμε λίγο την ψηφοφορία. Είστε έτοιμοι. Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία. Επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Για το ίδιο θέμα. Πέρασε τις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται 18 ψήφοι υπέρ, 1 κατά. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρέ δυσκολίε όσον αφορά τη χρηματοοικονομική του σταθερότητα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε για το σχέδιο ψηφίσματος. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Σημείο 7. Πρωτόκολλο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δημοκρατίας της Γκαμπών Σημείο υπαριθμών 7 της ημερήσιας διάταξης. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Έκανα λάθος εγώ. Με συγχωρείτε, ήμουν αφηρημένος. Ζητώ συγγνώμη. Ε, πάμε πάλι από την αρχή. Σημείο 6. Έκανε λάθος με τον κατάλογο ψηφοφορίας του προηγούμενου θέματος. Έκθεση της κυρίας Πατράων Νέβες χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά την χρηματοοικονομική του σταθερότητα. Ξεκινούμε λοιπόν τροπολογία υπαριθμών 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία τροπολογια υπεριθμών Άρχεται η ψηφοφορια περαση ψηφοφορία εγκρινεται Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Κυρία Λεβίν, παρακαλώ. Δεν βλέπουμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην οθόνη. Βάλε. Vale. No. Votamos entonces la 4. Comienza. Ωραία. Τέσσερα. Άρχεται η ψηφοφορία. Και αν ε, δεν το βλέπετε στην οθόνη θα σας το λέω εγώ. Πέρας τη ψηφοφορίας. Το βλέπετε. Μην το σβήνετε ακόμα. 16 ψήφοι υπέρ, 2 κατά, αν δεν κάνω λάθος. Τροπολογία υπαριθμών 4 και πάλι. Άρχεται η ψηφοφορία. Την 4 ψηφίζουμε. Πέρα τη ψηφοφορία. 15 υπέρ, 2 κατά ήταν. Λοιπόν, τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. 16 ψήφοι υπέρ, 3 κατά, εγκρίνεται. Τώρα φαίνεται και στην οθόνη. Τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η νομοθετική πρόταση ως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και το σχέδιο ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται 17 ψήφοι υπέρ, μία κατά, καμία αποχή. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Πρωτόκολλο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκαμπών. Έκθεση του κυρίου Φερέρα. Μία τροπολογία, ένα της κυρίας Πατράγου. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τι, όχι. Εγκρίνεται να ψηφίσουμε τώρα το ψήφισμα. Τροποποιηθέν. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται 18 υπέρ, ε, μία ψήφος κατά. Να περάσουμε στην επόμενη υγεία των ζώων. Γιατί το 8 αναβάλλεται. Τροπολογία 2 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 3 άρχεται. Κύριε Άγνιο. Ε, δεν ξέρω, είναι λίγο αργή η αγγλική μετάφραση. Ε, ε, δεν προλαβαίνω να ψηφίσω και λέτε ότι έχει λήξει η ψηφοφορία. Εντάξει, θα, θα σας δίνω λίγο περισσότερο χρόνο. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς ένα αριθμό ε, άρχεται πέρας. Εν πάση θα μιλάω πιο αργά. Λοιπόν, την τρία την ψηφίσαμε έτσι, η τροπολογία 4. Α, 3. 3, 3. Άρχεται. Λοιπόν, τέσσερα άρχεται. Ε, τρία λοιπόν. Τροπολογία αριθμός τρία άρχεται. Περάς. Εγκρίνεται. Τροπολογία τέσσερα άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 άρχεται πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 7. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 54. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. 11. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 55. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 56. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 57. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Λοιπόν, από κοινού. Από την 13 έως και την 16. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνονται. Μισό λεπτό, Α, δεν είχε μετρήσει η ψήφος του κυρίου Γκάλαχερ που είναι αρνητική. Οπότε νομίζω ότι υπήρχε ισοψηφία, οπότε θα απορρίπτονταν. Να ξανακάνουν ψηφοφορία των, 13, των τροπολογιών 13 έως 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 19 και ψήφος αρνητική του κυρίου Γκάλαχερ, οπότε απορρίπτονται. Οπότε, 13. 13 λοιπόν. Άρχεται. Πέρασε. Μισό λεπτό. Εάν ε, απορριφθούν από κοινού, απορρίπτονται όλες. Είναι σαφές. Λοιπόν, επειδή το ε, από κοινού απορρίφθηκαν, θα ψηφίσουμε μία-μία. Τροπολογία 13, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 11-9. 14, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 15, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 16. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα δεν καταλαβαίνω. Από κοινού απορρίφθηκαν και μία-μία εγκρίνονται. Είναι τα μυστήρια της Επιτροπής Αλίας. Καλά δεν πειράζει. Ε, εν πάση περιπτώσει. Εγκρίθηκαν τελικά, εντάξει, όλες. Λοιπόν, από κοινού 17 και 18. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνονται. Οπότε, οπότε, 19 έως 24 και 35. Ναι, ναι, ναι, μέτρησα και την ψήφο του κυρίου Γκάραχερ. 19 έως 24 και 35 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτονται. Οπότε, μία-μία τώρα, 19. πέρασε Εγκρίνεται. 20. Άρχεται. 20 ε, λέω. 20. Τροπολογία 20. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 21. Τι όχι. Η κυρία Λοβίν. Εμείς δεν ψηφίσαμε. Α, καλά, καλά. Να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Για την 20. Για την 20. Να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Εντάξει, εντάξει, ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 19. Ή 21. 21. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 22. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 23. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 24. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 35. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Μήπως θα πρέπει να κάνουμε καμιά μελέτη. Δεν έχει έννοια να ψηφίζουμε από κοινό τροπολογίες γιατί μετά τις ψηφίζουμε και μία-μία. Λοιπόν, όχι, την ψηφίσαμε 35. Την ψηφίσαμε λέω. Μα μόλις ψηφίσαμε 35. Λοιπόν, να ψηφίσουμε, να ξαναψηφίσουμε την 35. Γιατί μου είπανε ότι δεν την ψηφίσαμε. 35. Ας επαναλάβουμε την ψηφοφορία για την 35. Πέρας. Εγκρίνεται. 58. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 25 άρχεται πέρας φωνάζω πολύ και θα κουφάζουν τους, τους διερμηνείς εν πάση περιπτώσει άρχεται 26 συγγνώμη που το είπα καλά πέρας απορρίπτεται από κοινού 27-28 άρχεται πέρας Γκάλα χερκατά. Α, α, α, λειτουργεί η κάρτα, η κάρτα σας. Οπότε ε, συμπεριλαμβάνεται η ψήφο σας, οπότε εγκρίνονται. «29 με 34» λέει ο, ο Ha sido en bloque de 29 a 33. A ver si un poco. 34. 34. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ψηφίσαμε από την 29 στο 33 από κοινού. Α, συγγνώμη, 27-28. Τώρα ψη... ψηφίζουμε 29 έως 33. Άρχεται. Πέρασε εγκρίνονται. Οπότε περνάμε στη 34. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. 36. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. 37. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Από κοινού 38 έως και 43 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνονται. Από κοινού 44-45 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνονται. Από κοινού 46 με 51 άρχεται. Πέρασε. 46 με 51 εγκρίνονται. 52 άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται η 52. 53 άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται 13, 6 και μία αποχή. Ωραία. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο, 10. Πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών. Έκθεση, γνωμοδότηση μάλλον του κυρίου Ντέιβις. Τροπολογία 4. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 5. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 21 καταπίπτει. 22. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 23. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 6. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η 24 καταπίπτει. 8. Άρχεται. Την 8 λοιπόν άρχεται η ψηφοφορία το πρώτο τμήμα. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 29. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 15. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 8. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 25, όχι, καταπίπτει. 11. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Άρχεται. Πέρας Πέραση πληροφορία εγκρίνεται 26. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 14. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 27. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 28. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ένα. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεκαέξι. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Δύο. Πέρα. Πέρας. Εγκρίνεται. 17. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 18. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Πρώτο τμήμα της τροπολογίας παριθμών 3 που είναι πανομοιότυπο με το πρώτο τμήμα της 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας παριθμών 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και τώρα Τροπολογία 19, δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η γνωμοδότηση λοιπόν, όπως τροποποιήθηκε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας εγκρίνεται 13 ψήφοι υπέρ, 7 κατά. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο στην ημερησία διάταξη. Η απαλλαγή του 2012 για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλίας. Τροπολογία υπερθμών 1, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Τροπολογία 2, άρχεται η ψηφοφορία, Πέρας τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τη γνωμοδότηση λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας τη ψηφοφορίας. εγκρίνεται. 18 ψήφοι υπέρ, μία κατά και τέλος περνάμε στην ε, απαλλαγή 2012 για το Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δύο τροπολογίες, η ένα πρώτα, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Δεύτερη τροπολογία, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τη γνωμοδότηση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 18 ψήφοι υπέρ, μία κατά. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η ψηφοφορία. Πέρας λοιπόν της απόψινής συνεδρίασης και συνεχίζουμε με τη συνεδρίαση των συντονιστών. Ευχαριστώ λοιπόν τους υπολείπους, εσάβριον τα σπηδαία, στις 9 το πρωί στην αίθουσα της Επιτροπής Γυναικών. Σας υπενθυμίζω για να ψηφίσουμε εκεί.